πρόοδο του Κωσυφοπεδίου. Θα δώσω το λόγο ε, στην εκπρόσωπο πάλι του Συμβουλίου. Έχετε το μικρόφωνο. Αγαπητά μέλη, Πρόεδρε, Επίτροπε, να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την προσπάθειά της στο Κωσυφοπέδιο και να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο που μου δίνει την ευκαιρία να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του το Δεκέμβριο του 2014 σημείωσε την έναρξη τον μήνα Ιούλιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κοσφοπέδιο. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει τις απαιτούμενες προς υπογραφή προτάσεις το ταχύτερο δυνατόν. Το Συμβούλιο επίσης χαιρέτησε την υπερπίληση των εμποδίων που είχε προϋπάρξει. Ζητά από τις νέες αρχές της χώρας να αρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν τον διάλογο με, το, με την Σερβία. Ζητάμε από το Κοσφοπέδιο να συγκεντρώσει την προσοχή του στην εφαρμογή ενός συνολικού πακέτου μεταρρυθμιστικού υποχρεωτικού θα έλεγα στα πλαίσια της προτινόμενης συμφωνίας. Πρόοδος λοιπόν προς την ευρωπαϊκή οικογένεια είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα αυτή και τους πολίτες της. Οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου απαιτούν ε, να υπάρξουν το ταχύτερο δυνατόν αποτελέσματα. Απαιτείται λοιπόν σαφής πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στην βελτίωση του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και της εντατικοποίησης της καταπολέμησης ε, του εγκλήματος και της διαφθοράς. Η πρόοδος του κοσφοπεδίου μέχρι τώρα ήταν θετική αλλά επίσης υπενθυμίζουμε ότι το κοσυφοπέδιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα που ήρθαν στην επιφάνεια στα πλαίσια του διαλόγου για τις θεωρήσεις, ε, στα πλαίσια της ε, ε, μείωσης των κινδύνων που μπορεί να υπάρξουν εφόσον φιλελευθερωποιηθεί το καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων. Συνεπώς τα οικονομικά μέτρα και η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας είναι κάτι το απαραίτητο επιγόντως. Υπάρχουν προτεραιότητες και στον τομέα των εκλογικών μεταρρυθμίσεων και της προστασίας των μειονοτήτων. Η Επιτροπή για τα προγράμματα μεταρρύθμισης ε, θα έλεγα ε, καλύπτει πολλούς από τους στόχους στο κοσυφοπέδιο ελπίζουμε να βοηθήσει και την εφαρμογή του πακέτου οικονομικών μεταρρυθμίσεων της χώρας. Η διαδικασία εξομάλυνσης με την Σερβία, των σχέσεων με τη Σερβία, έχει σημειώσει πρόοδο σημαντική. Το κοσυφοπέδιο θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει έναν ενεργό και επικοδομητικό ρόλο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος και για τη Σερβία και το Κοσφοπέδιο. Συνεπώς η εξομάλυνση των σχέσεων είναι βασικός στόχος του Κοσφοπεδίου. Προς την κατεύθυνση αυτή επιτρέψτε μου να χαιρετήσω για μια ακόμη φορά την επανέναρξη του διαλόγου υψηλού επίπεδου της 9 Φεβρουαρίου ανάμεσα στις δύο χώρες και την ολοκληρωτική αν θέλετε διαμόρφωση της συμφωνίας για τη δικαιοσύνη στο Κοσφοπέδιο. Είναι θετικά βήματα για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας των Βρυξελών. Καλωσορίζουμε επίσης την συμφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Μουστάφα και τον Πρωθυπουργό Βούτσιτς που αποφάσισαν από κοινού να αντιμετωπίσουν περιφερειακά θέματα μεταξύ των οποίων και το οξυμένο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης από το το οποίο επίσης περιλαμβάνεται σαν πρόβλημα και στο δικό σας ψήφισμα. Το Συμβούλιο συνεπώς θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύναγκης τις προσπάθειες του Κωσυφοπέδιου προς μια απτή, ορατή και ταυτόχρονα βιώσιμη πρόοδο στον τομέα της εξημάλυνσης των σχέσεων με τη Σερβία πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι συμφωνίες που έγιναν μέχρι τώρα και πρέπει οι δύο χώρες αυτές να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή οδό. Είναι βασική αρχή της προτινόμενης συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η οποία θα ενισχύσει την εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ένωση και το Κοσμοπέδιο. Τέλος, το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με αποτελεσματικό και στενό τρόπο με τη Γιούλεξ και θα πρέπει να συνεισφέρει στην ανεμπόδιστη και πλήρη εκτέλεση των εντολών της Γιούλεξ που ανανεώθηκαν πρόσφατα. Το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει και τις ανηλυμένες πολιτικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων που θα ε, προέλθουν ε, μετά τα αποτελέσματα των ερευνών της ειδική ε, ερευνητικής ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάν, ο Επίτροπος Χάν. Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε και κύριοι βουλευτές, καλωσορίζω το σχέδιο ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή σωμάτι του κοσφοπεδίου. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμμερίζονται το ίδιο όραμα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για το κοσφοπέδιο. Ε, μα ευχαριστεί η υποστήριξη που δίνεται και θέλουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μα. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το Κοινοβούλιο και την εισηγήτρια κυρία Λούνα στου επόμενε μήνε για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή προοπτική του κοσμοπεδίου. Βάσει και του σχεδίου ψηφίσματος, την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Πρίστινα υπογράμισε την ανάγκη οικονομικών μεταρρυθμίσεων για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη, σε θέσεις εργασίας, σε επενδύσεις, στην εκπαίδευση και σε καλύτερες συνθήκες ε, διαβίωσης των πολιτών του Κωσυφοπηδίου. Αυτό καλύπτει, ε, απαιτεί την, ε, θα αντιμετωπίσει του τους λόγους της μετανάστευσης. Η έκθεση τον Οκτώβριο εντόπισε τους βασικούς τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το κοσφοπέδιο. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, το κράτος δικαίου, την ε, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Και οι τρεις πτυχές είναι ουσιώδους χαρακτήρα στους τομείς αυτούς και θα δώσουν πολιτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για τη χώρα. Τον Ιούλιο συμπληρώσαμε τις, ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Σύνδεσης ε, και Συνεργασίας και μονογραφήσαμε το κείμενο με το κοσφοπέδιο. Όπως ξέρετε, η συμφωνία αυτή είναι μόνο ενωσιακή, όχι μεικτή. Ωστόσο υπογραμμίζω ότι είναι και πλήρης και στεναρή, καλύπτοντας όλους τους βασικούς τομείς που καλύπτουν και οι άλλες ε, αντίστοιχες ε, συμφωνίες στην περιοχή. Όταν τεθούν σε ισχύ νομίζω ότι θα υπάρχουν πολύ λίγες πρακτικές δυσκολίες μεταξύ αυτής και άλλων. Μετά την μονογραφή της ε, συμφωνίας μεταφράζονται τα σχέδια της, ε, αποφάσεων του Συμβουλίου και θα είναι έτοιμα στο τέλος του μήνα θα ζητήσω από το Συμβούλιο να εγκρίνει το πακέτο, ε, από την Επιτροπή να υπογραμμίσει, να υποστηρίξει το πακέτο τον Απρίλιο και να το υποβάλουμε κατόπιν στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να μονογραφηθεί τον, την Άνοιξη και μόλις υπογραφεί από την κυρία και από την πλευρά του Κοσμοπεδίου θα υποβληθεί σε εσά. Το Κοινοβούλιο θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Αν θέλουμε η συμφωνία να υλοποιηθεί στις αρχές του 16 θα πρέπει να το χωρίσει γρήγορα η υλοποίηση. Είμαστε έτοιμοι βεβαίως να υποστηρίξουμε να δώσουμε υποστήριξη σε όλο τι χρειάζεται. Όταν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σύναψης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης λόγω του ότι είναι μόνο ενωσιακή συμφωνία δεν χρειάζεται κύρωση από πλευράς κρατών, άρα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα τεθεί σε άμεση ισχύ η συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας, κάτι που θα είναι ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί για πρώτη φορά θα υπάρξει συμβατική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου, η οποία παρέχει δικαιώματα σε, και υποχρεώσεις, ε, δικαιώματα και πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα και υποχρεώσεις. Και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε αυτό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση της θα είναι προς όφελος όλων. Προσβλέπω στην συνεχιζόμενη υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, δεν θα δεχθώ μπλε κάρτες. Θα δεχθώ όμως έξι συναδέλφους για ένα λεπτό τον καθένα. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο ομιλία σας. Κυρία Λούνατσικ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία ώστε να φτάσουμε σε ένα σε μεγάλο βαθμό συνενετικό κείμενο το οποίο ελπίζω ότι θα επιτύχει υψηλή πλειοψηφία αύριο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Κωσυφοπέδιο αναφέρθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως γιατί χιλιάδες ετούντες άσυλο ήρθαν από τη Σερβία και στη συνέχεια και στην, πέρασαν και στην Αυστρία και σε άλλες χώρες. Αυτό δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στο Κωσυφοπέδιο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ε, μειωθεί αυτή η κατάσταση, διότι στο Κωσυφοπέδιο πολλοί ότι οι βάση των υποσχέσεων που τους είχαν δοθεί είναι όντως ψευδέστηση. Οι αρχές και της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου προσπαθούν να εμποδίσουν τους εμπόρους ανθρώπων που τροφοδοτούν τέτοιες ψευδεστήσεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω και κάτι ακόμη. Στην έκθεση αυτή, όπως και σε πολλές άλλες πριν από αυτήν, ζητώ να δοθεί απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίου για το κωσυφοπέδιο το συντομότερο δυνατόν. Αν ήδη είχαμε την απελευθέρωση θεωρήσεων, δεν θα ένιωθαν κλειδωμένοι μέσα στη χώρα του. Θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε τρει μήνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γυρίσουν και δεν θα είχαν την εντύπωση ότι πρέπει να φύγουν γιατί διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν ποτέ. Χαίρομαι που πρόσφατα ο Επίτροπο Αβραμόπουλο είπε ότι το κοσυφοπαίδιο βρίσκεται στο τελευταίο τμήμα του δρόμου, τον οποίο διατρέχει και θα έχουμε σύντομα καλά νέα για το κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει να βελτιωθεί βεβαίως η κατάσταση ε, και για την ανεργία των νέων και να αντιμετωπίσουμε την διαφθορά. Η κυβέρνηση θα πρέπει να το κάνει αυτό ε, και να αντιμετωπίσει και ε, μέλη του κόμματος και πολλών θεσμών. Μετά από έξι μήνες ε, αδιεξόδου. Χαίρομαι που σχηματίστηκε πλέον κυβέρνηση με πολύ μικρή συμμετοχή γυναικών όμως. Ελπίζω ότι θα περάσει σύντομα μια νομοθεσία στο ειδικό δικαστήριο και εδώ δεν μιλάμε για τον KLA γενικά, μιλάμε για συγκεκριμένα μέλη του KLA που μπορεί να διέπραξαν κάποια εγκλήματα. Χαίρομαι που έχει ε, αναλυθεί εκ νέου διάλογος μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Υπάρχουν ακόμη θέματα που πρέπει να συζητηθούν βουλευτές του Κωσυφοπεδίου δεν επιτρέπεται ακόμη να συμμετέχουν σε πολλές συνεδριάσεις στα πλαίσια της ε, Κοινοβουλευτικής ε, Επιτροπής και επομένως είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακόμη, πέντε κράτη-μέλη ακόμη δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπαίδιο και αυτό εμποδίζει την πρόοδο και χαίρομαι που ακούω από τον Επίτροπο Χάν ότι η ε, συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης θα συζητηθεί σύντομα και ελπίζω να υπάρξει σημαντική πρόοδος. Διαβάστε το κείμενο παρακαλώ που μιλάει και για την EULEX και ε, για τις διατάξεις ε, σε σχέση με τη διαφθορά. Δεν θα πρέπει να παραμείνει οτιδήποτε θα δημιουργήσει προβλήματα στην αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ. Επόμενο ομιλητή ο κύριο Αντάκτουσον. Δεν τον βλέπω όμω στην αίθουσα. Θα περάσω στον κύριο Παντσέρη. Δύο λεπτά. E Ευχαριστώ για την δουλειά της κυρίας ε, Λούνατσεκ ε, που εδώ και χρόνια παρακολουθεί την πολιτική εξέλιξη στο Κωσφοπέδιο. Το ψήφισμα που έχει υποβληθεί είναι ισορροπημένο και δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Το κοσφοπέδιο, όπω αναφέρθηκε, είναι σε μια απόλυτα μεταβατική φάση και σίγουρα έχουμε θετική αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της πολιτικής αβεβαιότητας μετά την ε, διαμόρφωση νέας κυβέρνησης. Βέβαια υπάρχει και άλλος δρόμος τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις με αποφασιστικότητα, να ενισχυθεί με αποτελεσματικό τρόπο η σημασία της δικαιοσύνης και των νόμων και η αποκατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων. Επίσης σημαντικό είναι να ξεκινήσει και να, συνε... και να ολοκληρωθεί η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, ενώ πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική που αντιμετωπίζει την μεγάλη ανεργία των νέων ιδίως με οικονομικές, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Κατ' ουσία πρέπει να δοκιμάσουμε τη νέα κυβέρνηση μετρώντας τις ικανότητές της να εργάζεται προς όφελος των στόχων αυτών. Σίγουρα θα υπάρξει υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρότριση προς την κατεύθυνση αυτή γιατί οι στόχοι πρέπει να υλοποιηθούν. Ωστόσο παραμένουν κάποιες ανησυχίες που αφορούν στην ανεξαρτησία, την αξιοπιστία και την αμεροληψία των δικαστών και εισαγγελέων. Ε, μια λειτουργούσα δικαιοσύνη είναι βασικό στοιχείο μιας δημοκρατίας. Η αποστολή Έουλεξ είναι ένα θέμα που μας ενισχύει στο ψήφισμα, αναφέρεται η ανησυχία μας για κάποιες κατηγορίες διαφθοράς που θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Ένωσης. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε για να βοηθήσουμε το Κόσοβο να ε, γίνει πιο δημοκρατικό και να βοηθήσει στην σταθερότητα της περιοχής. Πιστεύω ότι το ψήφισμα προς την κατεύθυνση αυτή πηγαίνει. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κάρσκι. Πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε, το 2005 η γερμανική αντικατασκοπία αναφέρθηκε στο Κοσμοπέδιο ως ένα σοβαρό χώρο μαφίας που δημιουργεί προβλήματα σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε το, την εξαρτησία του Κοσμοπεδίου. Θέλω να επαναλάβω ότι τούτο ήταν τεράστιο πολιτικό και γεωπολιτικό λάθος. Οι αρχές και οι απαιτήσει της κρατικής υπόστασης δεν πληρούνται εκεί είναι μάλλον οργανώσεις εγκληματικές που δημιούργησαν μια ομάδα που δεν νομίζω ότι μπορεί να καλείται ως κράτος. Το κράτος κυριαρχείται από μαφίες που ε, αντλούν τους πόρους από την διακίνηση ε, ηρωίνης και ε, οργάνων, ανθρώπινων οργάνων. Ταυτόχρονα εμείς ε, διαπραγματευόμαστε με τη Σερβία και ταυτόχρονα με το κοσφοπέδιο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τις σχέσεις μας με τη Σερβία προς όφελος της Ρωσίας. ο Πούτιν θα είναι χαρούμενος στο να βοηθήσει να χάσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβία και αν χάσουμε τη Σερβία χάνουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων. Ο Επίτροπος ανέφερε και ένα άλλο θέμα. Ήδη αναγνωρίσαμε το ότι ε, δεν αναγνωρίσαμε το κράτος όλα τα, το κράτος Κωσοβίου, όλα τα κράτη της Ένωσης και προχωρούμε στη διαμόρφωση μιας μόνο ενωσιακής συμφωνίας και όχι μεικτής συμφωνίας. Και άλλο λάθος. Σας ευχαριστώ. Βάουτμαντς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βασικά την κυρία Λούνατσεκ για μια πράγματι εξαιρετική έκθεση. Ξέρετε ότι το Κωσυφοπέδιο είναι μια χώρα την οποία αγαπώ πολύ. Έχω πάει επανειλημμένα. Είχα συνοδεύσει και τον βασιλέα του Βελγίου εκεί και τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Γκί Φερχόφστατ είχα δει τις καταστροφές που είχε προκαλέσει ο πόλεμος στην χώρα αυτή και τελευταία φορά πήγα το 2014. Στα χαρτιά έχουν γίνει πολλά θετικά, αλλά στην πρακτική πολλά μένει να γίνουν. Οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας φυσικά τις προσπάθειες των κατοίκων της χώρας, αλλά δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε και τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν. Πιστεύω και η πολιτική μου ομάδα ότι το κοσυφοπέδιο κάποια στιγμή θα πρέπει να τύχει αναγνώρισης από το σύνολο των υπολείπων χωρών. Είναι μία από τις πιο φτωχές και πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης με ανεργία 35%. Η Πρίστινα λοιπόν έχει ανάγκη από την Ευρώπη για να βελτιωθεί η κατάσταση σε επίπεδο κράτους δικαίου, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και εξόδου των κατοίκων. Ε, ξέρουμε ότι τους τρεις τελευταίους μήνες έχουν φύγει 35.000 ε, κάτοικοι της χώρας αυτής. Αυτή είναι απίστευτη αριθμή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν αλλαγές στη χώρα αυτή και σε οικονομικό επίπεδο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να γεννήσουν θέσεις απασχόλησης και να λειτουργήσει σαν βιώσιμη χώρα το κοσυφοπέδιο. Για ένα λεπτό ο κύριος Χρυσόγονος. It's late. I should be forgiven. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 16 χρόνια ένας αριθμός κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη ΣΥΠΑ αποφάσισαν να καταπατήσουν την αρχή της μη αλλαγής συνόρων στην ευρώπη και να αποσπάσουν με τη βία ένα μέρος της σερβικής επικράτειας για να το μετατρέψουν σε προτεκτοράτο. από τότε η διοίκηση του κωσυφοπεδίου έχει αποδειχθεί διαρκής ευρωπαϊκή αποτυχία η οποία διαφαίνεται και από την τελευταία έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής. το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής αυξάνεται αλλά η αύξηση διοχετεύεται στο οργανωμένο έγκλημα ενώ η εξαθλίωση των ανθρώπων ολοένα επιδεινώνεται και δημιουργεί κύμα φυγής προς την ευρώπη με αποτέλεσμα ο πληθυσμός από δύο εκατομμύρια το 2009 να έχει πέσει στο ένα εκατομμύριο το 2012. Οι εξαγωγές είναι πρακτικά ανύπαρκτες, η ανεργία παρά τη μετανάστευση βρίσκεται στο 30% και η διαφθορά κυριαρχεί. Η Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει την αποτυχία της και να περιορίσει την ανάμειξή της στο Κωσφοπέδιο. περισσότερη ζημιά κάνουμε εκεί παρά όφελος. οι κάτοικοι του Κωσφοπέδιου έχουν μια πολύ δύσκολη θα έλεγα κατάσταση μπροστά τους. Στην ουσία ακόμα όπως είπε και ένας γνωστός διανοούμενος και καλλιτέχνης η μόνη λύση για αυτούς ε, είναι η μαύρη οικονομία και η μετανάστευση. Ένας λοιπόν στους τρεις κατοίκους της χώρας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ένας από τους τρεις δεν έχει δουλειά. Πρέπει λοιπόν ε, να εξηγήσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι τον τελευταίο καιρό 18.000 κάτοικοι της χώρας αυτής πήγαν στη Γερμανία Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με το οργανωμένο έγκλημα, σωματεμπορία, ε, εμπορία ε, γενικά ε, απαγορευμένων ουσιών κτλ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να βγει από την κρίση. Αν δεν βοηθήσουμε τη χώρα αυτή τότε δεν μπορεί να στρέψει με αισιοδοξία το βλέμμα στο μέλλον. Η έκθεση της κυρίας Λούνατσεκ είναι μια καλή προσπάθεια και η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο θα πρέπει να συνεχίσουν παράλληλα την πορεία προς την ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορφάι, αλλά η κυρία Μορφάι δεν είναι στην Ολομέλεια και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για ένα λεπτό. Στον κύριο Μακάλιστερ, συγγνώμη, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από τρει εβδομάδε πήγα στο Κωσυφοπαίδιο και μεταξύ άλλων συνομίλησα και με τον Πρωθυπουργό, κύριο Μουσταφά. Και το θέμα ήταν η έκθεση προόδου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ω εισηγήτρια. Ένα βασικό θέμα στην Πρίστινα ήταν το κύμα ετούντων άσυλο από το Κωσυφοπαίδιο που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρθηκε και σήμερα. Και η Γερμανία θίγεται ιδιαίτερα από αυτό το κύμα. Πρώτο σημαντικό μέτρο πρόσθετη έλεγχη στα σύνορα που φαίνεται να οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη επιτυχία. Χρησιμοποιώ την ευκαιρία διότι σήμερα παρακολουθεί τη συζήτηση και ο πρέσβης ε, του Κοσμοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, πολύ σημαντική η εκστρατεία ενημέρωση επιτόπου, δηλαδή ότι το Κοσμοπέδιο είναι μια ασφαλής χώρα προέλευσης. Δεν έχουν δηλαδή καμία πιθανότητα αναγνώρισης ε, τον άσυλο στη Γερμανία όσοι ζητούν άσυλο από το Κοσμοπέδιο. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει αυτή η εκστρατεία ενημέρωση επιτόπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σε κάθε πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό. Ο κ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το 2014 ήταν μια σημαντική χρονιά για το κοσμοπέδιο και την διαδικασία προσέγγιση του προ την Ένωση. Η υπογραφή τη Συμφωνία Σύνδεση και Σταθεροποίηση ανοίγει την δυνατότητα ενιαίου οικονομικού χώρου. Δεν πρέπει να σταματήσουμε ωστόσο μόνο εκεί, αλλά να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενό πλήρου χώρου ενιαία αγορά με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και από την άποψη το 2014 ήταν σημαντικό. Το, η κυβέρνηση διαμόρφωσε μια συμβουλευτική ομάδα για τα ε, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και των ΛΟΑΤ, ενώ ταυτόχρονα ε, υιοθέτησε την παγκόσμια ρύθμιση για την ε, αντιμετώπιση της ομοφιλοφοβίας. Δεν υπήρξαν ωστόσο επεισόδια ε, όπου τον, υπήρξαν περιπτώσεις όπου εμφανίστηκαν σε κάποιες περιοχές και η σημαία με το ουράνιο τόξο. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Λούνατσεκ για την εξαιρετική έκθεσή της που θα υπερψηφίσω αύριο στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζαμπάσκι για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Συνάδελφοι, να συγχαρώ καταρχάς την κυρία Λούνατσεκ. Μπράβο της για την πολύ καλή έκθεση. Ήταν πολλή δουλειά. Ήμουν σκιώδης εισηγητής και νομίζω ότι το κείμενο καλύπτει πολλά από αυτά που είπαμε και αντιμετωπίζει πολλές από τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να αναφέρουμε το θέμα των κατηγοριών για τη διαφθορά στα πλαίσια της Ulex. Επίσης, το θέμα της διακίνησης ναρκωτικών, άλλα σοβαρά εγκλήματα. Αυτό που με ανησυχεί πάνω απ' όλα ωστόσο είναι το ότι στο Κοσφοπέδιο υπάρχουν ξένοι μαχητές που έρχονται στην Ευρώπη. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο κύριος Κούτσακ για ένα λεπτό. Ο Κούκαν. Πρόεδρε. Επίτροπε. Υπουργέ. Το 2014 ήταν σημαντική χρονιά για την ενταξιακή προοπτική του Κοσποβιδίου με την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθερότητας που ελπίζουμε να υλοποιηθεί την άνοιξη, αυτή την άνοιξη. Έγιναν εκλογές. Οι διεθνείς παρατηρητές είπαν όλοι πως ήταν δημοκρατικές και με διαφάνεια. Παρά τις δυσκολίες του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων κομμάτων που κράτησαν 6 μήνες, τώρα έχουμε κυβέρνηση. Το Κωσοβό πρέπει να συνεχίσει τις βασικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του οικονομικού ε, περιβάλλοντος. Τα ζητήματα τα βασικά αφορούν τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, το οργανωμένο έγκλημα, την διαφθορά. Πρέπει να ξεκινήσουν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να χτυπήσουμε την ε, ανεργία. Γι' αυτό το Συμβούλιο πρέπει να, υπογραμμίσει, να υπογράψει την συμφωνία και να συμπεριλάβει στα ευρωπαϊκά προγράμματα το Κωσοβέδου κάτι που βοηθήσει την οικονομία της χώρας και την ε, συνεργασία της με σε διαφορε τομεί. Ο κύριος Στρέκες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντίθετα με την εποχή της εφορίας μετά την ανεξαρτησία, είναι ανησυχητική η τωρινή κατάσταση. Η ένδια, η ανεργία, η εσωτερική κατάσταση ταραχές στις οποίες οι πολίτες αυτού του νέου κράτους δεν μπορούν να χαρούν την ελευθερία ή την ανεξαρτησία τους ε, ή την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και προτιμούν να μεταναστεύουν κατά χιλιάδες. Κυρίως ευθύνεται η ε, πολιτική η εσωτερική πολιτική τάξη Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το κοσυφοπαίδιο σε αυτή την ε, κρίση που οξύνεται. Η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα στο κοσυφοπαίδιο. Εκεί πρέπει να αντιμετωπίσουν την πηγή των κυμάτων μετανάστευσης. Και η Σερβία δεν θα πρέπει να θέτει εμπόδια, θα πρέπει όμως ε, να βοηθά την πρώην επαρχία της στην ανάπτυξή της. Ευχαριστούμε και δίνω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Μόλνα. Κύριε Πρόεδρε, το 2008 η Ευρώπη έδωσε τη δυνατότητα στο Κωσυφοπαίδιο να διακήρυξει την ανεξαρτησία του και ξεκίνησε και η ειρηνευτική διαδικασία στα Βαλκάνια. Τώρα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μεταναστευτικά κύματα του 2014 δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει τη χώρα του για να περάσει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Πώς είναι, δυτικό, είναι δυνατόν αυτό. Οι κατοίκοι του Κωσυφοπεδίου έχουν δύο επιλογές. Είτε να αντέξουν τη φτώχεια στη χώρα τους ή να προσπαθήσουν να φύγουν και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για όλους τους κατοίκους του Κωσυφοπεδίου και αυτούς που μένουν στη χώρα τους και αυτούς που έρχονται στην Ευρώπη. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε εξτρεμιστικά κόμματα τα οποία κεφαλαιοποιούν αυτά τα πολιτικά ζητήματα. Μερικές φορές ακόμη και κυβερνητικά κόμματα μιλούν για αυτούς τους μετανάστες ως οικονομικούς μετανάστες. Η Ευρώπη έχει πολλή δουλειά να κάνει και τα κράτη-μέλη έχουν πολλά να κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχατε ένα λεπτό και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την έκθεσή της και να την ευχαριστήσω για την προσπάθεια που καταβάλει για το κοσυφοπαίδιο. Μετά την, το διάστημα που πέρασε μετά τις εκλογές, η νέα κυβέρνηση του κοσυφοπαιδίου θα πρέπει να επικεντρωθεί σε βασικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της χώρας. Είναι σαφείς οι συνέπειες της αποτυχίας της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Το κοσυχοπαίδιο πρέπει να αντιμετωπίσει επιγόντως τα θέματα οικονομικής ανάπτυξης και το πρόβλημα της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας. Η, άνοδος, ε, η αύξηση των ετούντων άσυλο είναι μία μόνο από τις συνέπειες. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και να προχωρήσουμε ε, στα θέματα της απελευθέρωσης θεωρήσεων διαβατηρίου. Από την άλλη πλευρά, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Περιμένουμε επίσης και τα αποτελέσματα ερευνών ε, για θέματα διαφθοράς σε σχέση με την ε, EULEX. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας, πράγμα το οποίο και βεβαίως θέλουμε, θα πρέπει να χυθεί το φως σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράτη και ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ για την ισορροπημένη έκθεσή της καλωσορίζω την τελευταία πρόταση του Επιτρόπου Χάν. Η διαδικασία παρέχει υποσχέσεις. Στη συζήτηση μιλήσαμε για πολλά προβλήματα, ελλείψεις, ζητήματα. Κάποιοι μίλησαν για αρνητικές εξελίξεις στη χώρα. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προοπτικής, η έλλειψη ευκαιριών. Τι ευκαιρίες έχουν σε αυτό το πολύ μικρό κράτος που είναι. Τι συζητούμε όταν μιλούμε για τη δυνατότητα σύνδεσης ή προσχώρησης. Είναι να τους δώσουμε μία προοπτική και νομίζω ότι αυτή την προοπτική την χρωστάμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εμπειρία που είχε ολόκληρη αυτή η περιοχή. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κ. Μπόγκοβιτς, ένα λεπτό. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτούς που συνεχάρισαν την κυρία Λούνατσεκ. Εξαιρετική έκθεση. Μας δείχνει με πολύ σωστό τρόπο την κατάσταση στη χώρα αυτή. Συζητήσαμε τα του Κοσφοπεδίου και όταν συζητούσαμε ε, για τη Σερβία είπαμε ότι ήταν καλή και εκείνη η έκθεση όπως είναι και αυτή εδώ. Υπογραμμίζουν κάποια κομβικά προβλήματα που έχει η χώρα να αντιμετωπίσει όπως ε, το οργανωμένο έγκλημα, το θέμα των προσφύγων που αναζητούν το μέλλον τους και σε άλλες περιοχές, το τρομακτικό πρόβλημα της ανεργίας και θα συμφωνήσω με αυτούς οι οποίοι ε, υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η σωστή συνεργασία του Κωσφοπεδίου με τη Σερβία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, Φροντσούλιτσα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έγιναν βήματα, πρέπει όμως να υπάρξουν περισσότερα. Ιδιαίτερα για να βοηθήσουμε τη δικαστική εξουσία να πολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, να προωθήσουμε την απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια και την αηφορία ενεργειακά της χώρας. Απαιτείται επίσης η βελτίωση του ρόλου των γυναικών στην κυβέρνηση, και η προστασία της ελεύθερης έκφρασης. Εμείς παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις διαπραγματεύσεις Σερβίας Κοσφοπεδίου και θα ενισχύσουμε την συνεργασία μας με τη χώρα αυτή και στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να τεθεί το θέμα της Γιούλεξ, να δούμε αν πράγματι η Γιούλεξ λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ο κύριος Μωράης, ένα λεπτό. Ισλαμικών στοιχείων στο Κόσοβο δημιουργεί έντονες ανησυχίε στην περιοχή. Ήδη έχουν γίνει μαζικές συλλήψει υπόπτων για συμμετοχή σε πολεμικέ επιχειρήσεις στο Ιράκ και στη Συρία. Προβληματικό είναι επίσης και ο ρόλος συγκεκριμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων με προέλευση από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ τα αυξημένα μεταναστευτικά κύματα από το κόσοβο σε χώρες της ένωσης με πολυπληθείς αλβανικές μειονότητες εντείνουν την ανησυχία των πολιτών της ένωσης. ταυτόχρονα η αναβίωση του αλβανικού εθνικισμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς τα τύρανα προωθούν με μοχλό το κόσοβο την αλυτρωτική ιδέα της μεγάλης αλβανίας που διεκδικεί αλλαγή συνόρων στα βαλκάνια και εδάφη τα οποία ανήκουν στην ελλάδα. τέλος κυρία πρόεδρε διερωτώ πώς μπορεί να γίνει κάποτε μέλος ενδεχόμενα της ευρωπαϊκής ένωσης το κόσοβο από τη στιγμή που πέντε κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης δεν αναγνωρίζουν καν το κόσοβο ως κρατική οντότητα. ευχαριστώ. Το κοσίφο πέδιο χρειάζεται πολλέ μεταρρυθμίσει. Θέλουμε να το υποστηρίξουμε στον ευρωπαϊκό δρόμο του, αλλά είναι αναγκαίε οι μεταρρυθμίσει. Να τονίσω ιδίω κάτι που κανεί δεν ανάφερε μέχρι τώρα, την ανάγκη να προστατευτεί, να προστατευτούν τα δικαιώματα τη σερβική κοινότητα στο κοσμοπέδιο. Εγώ υποστηρίζω το υποστήριζα πάντα τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των Σέρβων στην Κροατία για παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία του σερβικής μειονότητας στο Κοσμοπέδιο. Μιλάμε για το μέλλον των Βαλκανίων εδώ. Μιλήσαμε για το μέλλον των Βαλκανίων ε, σήμερα το βράδυ από πολλούς τρόπους. Κάποια στιγμή ωστόσο ένα όραμα είναι να ενταχθεί όλη η Βαλκανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτή είναι η μόνη ουσιαστική προοπτική τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ε, το δικό μου παρελθόν ε, ε, Ρωμά θέλω να μιλήσω κατά των διακρίσεων κατά της μειονότητας των Ρωμά στο Κωσυφοπαίδιο σε θέματα που αφορούν την παιδεία, την στέγαση, την απασχόληση και την ύπαρξη ευκαιριών. Η μειονότητα των Ρωμά κινείται προς δυσμάς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια διακριτική μεταχείριση που δεν είναι αποδεκτή. Θα πρέπει η κοινότητα των Ρωμά να μπορεί να επιλέξει τη χώρα της αρεσκίας της. Υπάρχει μια προοπτική και αν ε, έχουν ε, περισσότερες δυνατότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έρθουν περισσότεροι στο Ηνωμένο Βασίλειο πράγμα το οποίο θα οδηγήσει ακόμη μεγαλύτερο κύμα δυσφορίας προς τους Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ομιλητή ο κ. Κορέο. Ένα λεπτό. Κ. Κοράο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ. Είναι επικοδομητική η έκθεσή της. Μιλήσαμε και για άλλες χώρες προηγουμένως και τώρα έχουμε την πιο δύσκολη περίπτωση. Είναι μια νέα χώρα, μια χώρα που δεν αναγνωρίζεται από πέντε χώρες της Ένωσης και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνει πολύ βιαστικά και να καθυστερήσει τις διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια φυσική διαδικασία προσέγγισης των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και πρέπει να τα δούμε ε, το μέλλον των σχέσεων της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση με επικοδομητικό τρόπο. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χάν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας προς τις πρωτοβουλίες μας στο Κοσμοπέδιο. Το σχέδιο ψηφίσματος που συζητήσατε τώρα είναι πολύ επικοδομητικό και ευχαριστώ την κυρία Ρούνατσεκ για την δουλειά που έκανε. Δύσκολη φαντάζομαι. Επίσης, δείχνει τη σημασία του κοσμοπεδίου για θέματα οικονομίας και κατά δικαίου αλλά δείχνει και το δρόμο προς εμπρός. Η σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα δώσει ενθαρρυντικά μηνύματα σε όλους τους πολίτες της χώρας, ε, τονίζοντας ότι το μέλλον της χώρας ε, έγκυται στην προσέγγιση της ε, με την Ευρώπη. Η ενταξιακή προοπτική είναι μεγάλο κίνητρο και για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων του κοσυφοπεδίου. Θέλω ωστόσο να ευχαριστήσω και παρουσία της πρέσβεως ε, όλες τις αρχές της χώρας, ιδίως το γραφείο του Πρωθυπουργού για την άμεση, γρήγορη και άμεση αντίδραση στο θέμα της ε, μεταναστευτικής ζωής που αντιμετωπίσαμε πέρυσι γιατί πέρασαν στους πολίτες της χώρας ότι δεν έχει νόημα να φύγουν από τη χώρα και να ζητήσουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν, νομίζω, σε σημαντική μείωση του αριθμού των μεταναστών, κάτι που είναι θετικό για την ποιότητα της διοίκησης και των πολιτικών στη χώρα. Ευχαριστώ και παρακαλώ να επιβάσετε τις ευχαριστίες μας στις αρχές της χώρας σας. Ίσως να μπορέσω να το κάνω κι εγώ, διότι σε δύο εβδομάδες θα βρεθώ στο, στη χώρα σας για να μετάσχω στην διάσκεψη των έξι των Δυτικών Βαλκανίων για θέματα διευκόλυνσης των μεταφορών όπου το κοσφοπέδιο μετέχει πλήρως σε όλες τις δραστηριότητες της περιοχής, προσπαθώντας να βελτιώσει την επικοινωνία την... μεταξύ των χωρών της περιοχής, βοηθώντας την αύξηση στην ανάπτυξη, την ευημερία της θέσης εργασία στην περιοχή. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για το Σουαπέδο και ευχαριστώ τους βουλευτές για την επικοδομητική δουλειά τους προς όφελος του Κωσυφοπεδίου και άρα και της Ευρώπης ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Τελευταία λέξη, η Υφυπουργό της Λετωνίας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βοηθά το κοσυφοπαίδιο Βασική ευθύνη όμως για την πρόοδο της χώρας ανήκει στους κατοίκους της χώρας αυτής, την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει την σημασία ολοκλήρωσης της Συμφωνίας Σύνδεσης το ταχύτερο δυνατόν. Θα είναι και μια σημαντική συνεισφορά στην περιφερειακή συνεργασία και σταθεροποίηση. θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω κίνητρα για μεταρρυθμίσεις στο Πέδιο. Περιμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Συμβούλιο πριν συνεχίσουμε. Θα εκδώσουμε μία απόφαση για να υπάρξει συμφωνία χωρίς καθυστέρηση. Οι μεταρρυθμίσεις είναι κρίσιμες και απαιτείται οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το καλό της χώρας και των πολιτών της. Οι μεταρρυθμίσεις είναι βασικές όχι για να κολακέψουν την Ένωση αλλά γιατί αυτές έχουν μεγάλη σημασία και είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμη φορά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ υπουργέ. Τελειώνει λοιπόν εδώ η συζήτηση. Υπάρχει μια πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ψηφίσουμε αύριο.